Καλημέρα σας. Θα αρχίσουμε επίσημα τώρα. Καλημέρα σας λέω. Πρώτο περάσουμε στην εξέταση μερισσίας διάταξης. Θα ήθελα, μια που δυστυχώς το ξεχνάω πάντα, θα ήθελα σήμερα να ευχαριστήσω τους διερμηνείς που είναι πάλι πολύ άριθμοι Σχεδόν πλήρες είναι η παρουσία τους. Όλες οι καμπίνες ερμηνείας είναι γεμάτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε και υποστηρίζετε την εργασία μας κατά τέτοιο καταπληκτικό τρόπο. Συνήθω ξεχνάμε να το πούμε. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι εξ όλων εκφράζομαι εδώ. <laughs> Παρατηρήστε εκτός μικροφόνου, δυστυχώς. Σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Εκτός από τα πρακτικά των περσμένων συνεδριάσεων μας που πρέπει να εγκρίνουμε, που νομίζω μπορούμε να το κάνουμε εδώ, δεν... νομίζω ότι υπάρχουν συμπληρωματικές παρατηρήσεις. Και μετά Έχουμε δύο πράγματα κατά νου για σήμερα. Καταρχήν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων πάνω στις παλιάριθμες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και έχω να πω εδώ κάτι δεν πρέπει να κάνουμε αυτό που γίνεται συνήθως δηλαδή συμφωνήσαμε σε συνομιλίες με τους συντονιστές τους και όδης εισηγητές κατόπιν βέβαια προτάσεως των εισηγητών, ότι θα ακολουθήσουμε διαφορετική από τη συνήθεια. και μετά η συγγήτρια υπάρχει ένα πρόβλημα, υπήρξε ένα τεχνικό, μια τεχνική διακοπή, πολύ σύντομη. Französisch geht nicht. Γαλλικά δεν ακούτε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Geht? Doch, hinten geht's. Peut-être tu... Sie telefonieren. Okay, I, I, I switch to English then if, if French is, is right. It's okay? Είναι εντάξει τώρα. Α, ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι συμφωνήσαμε με, τους, με την εισηγήτρια και τους κοιόδες εισηγητές και τους συντονιστές ότι η Περβόν Σπεχές είχε συμφωνήσει μέχρι τα τέλη του μηνός να εξετάσει την έκθεση και να υποβάλει μια νέα έκδοχη. Οι τροπολογίες που υπάρχουν και που υπάρχουν επιτάπητος τα προετοίμαζε ε, συμβαστικές τροπολογίες äh, και μέχρι την 31η Αυγούστου θα υπάρχει μια έκτακτη συνεδρία πάνω στο οποίο θα συζητηθούν αυτά τα ε, σημεία και ελπίζουμε αρχές Σεπτεμβρίου να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα και να μπορέσουμε έτσι να εγκρίνουμε τη νέα έκθεση με μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια. Στις 21 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή θα ψηφίσουμε πάνω σε αυτό και ελπίζω έτσι η ομάδα εργασίας, η έκτακτη ομάδα εργασίας του Προέδρου Φανερόπόη θα μπορέσει να παρουσιάσει τις προτάσεις της και θα θέλουμε να μπορούμε να συνεργαστούμε. Έχει αλλάξει λοιπόν κάπως η διαδικασία και γι' αυτό δεν θα περάσουμε σήμερα στην επιμέρους συζήτηση των 1.700 τροπολογιών äh, äh, αλλά θα ζητήσω από τους εκπροσώπου των πολιτικών ομάδων να κάνουν εισαγωγικά κάποια σύντομη äh, το άλλο είναι ότι όπως ξέρετε Γίνονται τεχνικές διακοπές. Apparently we have, we are, apparently we're having problems here with the, with the, with the technic, technical equipment, so... Θα συνεχίσω στα αγγλικά. Είναι ίσως τα πιο εύκολο για όλους. Να μπορούν όλοι να παρακολουθήσουν. As you know, as you know, the, the, Όπως ξέρετε, η Επιτροπή μας η έκτακτη επιτροπή κρίση έχει παρατοθεί στη λειτουργία της μέχρι του χρόνου του καλοκαίρι. Έτσι, η τελική έκθεση, γιατί αυτό που συζητάμε είναι η διάμεση έκθεση. Η τελική έκθεση θα ψηφιστεί στην ε, ε, Ολομέλεια του χρόνου τον Ιούλιο. Και θα πρέπει να έχουμε ψηφίσει εμείς στην Επιτροπή μας τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα Δηλαδή, λίγο πολύ θα έχουμε έξι μήνες για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Θα δούμε ποιο θα είναι το επίκεντρο των εργασιών αυτών. Και εδώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε το εξή, κυρίως οι και σκιώδεις εισηγητές, αλλά όλα τα μέλη. Να σκεφτείτε αυτοί οι επιπλέον έξι μήνες που θα έχουμε στη διάθεσή μας, ποιο θέμα θα πρέπει να έχουν έτσι ώστε το Σεπτέμβριο να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε πάνω σε ένα πρόγραμμα εργασίας για το υπόλοιπο του χρόνου ύπαρξης της Επιτροπής. Τούτο λεχθέντος. Θα ήθελα να καλέσω τώρα τα μέλη των πολιτικών ομάδων να σχολιάσουν. και προηγουμένω ίσω Περές να μας κάνει μια παρουσίαση και μετά θα περάσουν στους άλλους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτή την περιγραφή των σημείων για τις συζητήσεις μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που είναι παρόντες εδώ και όλους όσους έχουν συμβάλει με τις 1625 τροπολογίες που έχουν υποβληθεί ε, που δείχνει τη σπουδαιότητα αυτής της συζήτησης για μας για την προσθέμενη αξία πολλών από αυτές τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, διότι πιστεύω ότι στο περιεχόμενο των τροπολογιών υπάρχουν κάποιες, κάποια σημεία διαφωνίων, αλλά υπάρχουν και πολλά σημεία προσθέμενης αξίας. Και θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον καθένα γι' αυτό. Θα ήθελα να πω ε, σαφέστατα στον κάθε συνάδελφο ότι το σύνολο των 1.625 τροπολογιών έχουν αναγνωστεί και αναλυθεί μία-μία και όχι ε, όλη, η ουσία αυτών των τροπολογιών ε, θα εξαχθεί. Όταν βλέπω το περιεχόμενο των τροπολογιών, βλέπουμε ότι υπάρχουν μερικές φορές μέσα σε μια ομάδα συζητήσεις που δεν έχουν ακόμη ε, ολοκληρωθεί και δεν έχει ληφθεί απόφαση. Και θα πρέπει να σας υποδείξω ότι ίσως ε, λόγω ε, διανοητικής ειλικρίνειας όταν υποβάλλονται διάφορες τροπολογίες από, τους, από διάφορους συγγραφείς ε, διαφορετικών ομάδων πολλές φορές υπάρχει μία τροπολογία που φαίνεται να είναι η θέση της ομάδας και όχι οι μεμονωμένες θέσεις του ενός του άλλου κράτους μέλους. Ε, θα πρέπει να δώσουμε σημασία στην τροπολογία που έχει υποβληθεί από αυτό που φαίνεται, διαφαίνεται ως τοποθέτηση της ομάδας και όχι με μονομένη τοποθέτηση, αν είναι πολύ αντιφατικές μεταξύ τους. Κάτι άλλο μια τεχνική παρατήρηση. Έχουμε όλοι πει ότι αυτή η, ε, αυτή η έκθεση θα πρέπει να είναι εστιασμένη και να μην είναι πολύ μακροσκελής. Αλλά πρέπει να σας πω ότι εδώ δυσκολεύομαι διότι από το σύνολο των τροπολογιών που έχω λάβει έχω 410 ε, τροπολογίες ε, που αφορούν 168 παραγράφους, αλλά έχω 422 προτάσεις προσθήκης κειμένου. Ε, ακόμη και αν δεχτώ όλες τις τοπολογίες αφαίρεσης προσθήκης, θα καταλήξουμε σε μια πολύ πιο μακροσκελή έκθεση από αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, θα πρέπει να βρούμε μια χρυσή τομή ανάμεσα σε όλα αυτά τα σημεία. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι από, ε, ανάμεσα σε τρία ε, θέματα, η συνοχή, ε, μικρομεσαίες και εποπτεία, υπάρχουν πάρα πολλέ προσθέμενες προτάσει. Αντιλαμβάνουμε ότι είναι σημεία στα οποία τα μέλη θέλουν να δείξουμε περισσότερη εξειδίκευση, να εξειδικευτούμε περισσότερο. Και ε, προτείνω λοιπόν να συμπληρώσουμε την έκθεση προσθετοντα δύο ή τρεις παραγράφους στο κάθε ένα από αυτά τα σημεία. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει και εκεί να προσπαθήσουμε να ε, συρρυκνώσουμε λίγο το ε, κείμενο σε σχέση με όλε τι παραγράφου που προτείνονται ως προσθήκες σε αυτά τα τρία θέματα. Συνοχή, εποπτεία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, στην ουσία της συζήτησής μας, έχω, και έχω διαπιστώσει εδώ ότι ε, είναι αυτά τα σημεία διαφωνίας. Υπάρχει ένα λεκτικό ή διατυπώσεις που μπορεί να αμφισβητήσει κανείς και ο καθένας βέβαια θα πρότεινα κάτι που θα ε, επιτρέψει στον καθένα να συμφωνήσει ε, σε ένα κοινό λεκτικό. Όμως υπάρχουν και πιο δύσκολα σημεία και είναι ίσως σημεία τα οποία θα παραμείνουν ανοιχτά για διαπραγμάτευση ανάμεσά μας μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Και θα ήθελα εδώ να υποφεληθώ αυτή τη ανταλλαγή απόψεων για να τα αναφέρω. Υπάρχουν αρκετά, ε, με συγχωρείτε γι' αυτό, θα χρειαστεί να κάνω αυτή την παρουσίαση πρωτού μπούμε στη συζήτηση. Στην παράγραφο 20 που αφορά το ιστορικό πλαίσιο που εντοπίζει την φύση της κρίσης την οποία διατρέχουμε, ε, νομίζω είναι χρήσιμο να εντοπίσουμε αυτά τα ιστορικά γεγονότα, τα στοιχεία του πλαισίου του γενικού, αλλά υπάρχουν και σημεία διαφωνίας ε, σχετικά με την αναφορά της ρήξης στο οικονομικό σύστημα, το παγκόσμιο, που αποτελεί το, το Bretton Woods, το σύστημα Bretton Woods. Εδώ νομίζω υπάρχει ένα σημείο το οποίο θα συζητηθεί. Τώρα, παράγραφος, δεν ξέρω αν έχω δει στην έκθεση, προσπαθώ να ακολουθήσω την έκθεση. 120 παράγραφος που αποτελεί την ισχυρή πρόταση στο θέμα της ενέργειας. Εδώ υπάρχουν προτάσεις αφαίρεσης ε, από τους ελεύθερους και από την ομάδα του ΕΛΚ. Έχω διάφορα ερωτηματικά και κάποια επιχειρηματολογία εδώ για τα... Ε, το ερώτημα είναι μήπως υπάρχει διαφωνία στην ουσία της πρότασης ή, ή μήπως είναι μια προ... Ε, το ερώτημα είναι ότι είναι μια πρόταση εκτός θέματος σε ό,τι αφορά το διακύβευμα της πρότασης. Εγώ πιστεύω πιο πολύ ότι είναι ένα πρόβλημα ουσίας. Διότι στην πραγματικότητα η συγκεκριμένη εφαρμογή της πρότασης, όπως φαίνεται στην παράγραφο 120, ε, ε, περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 122. Εκεί δεν υπάρχει αμφισβήτηση, υπάρχει λιγότερη αμφισβήτηση. Άρα, αναρωτιέμαι ειλικρινά εδώ, αν μπορούμε να βρούμε μία συμφωνία στην παράγραφο 120. Γιατί διότι υπάρχει ένα ολόκληρο διακύβευμα που είναι στην αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση συστάθηκε με βάση τον άνθρακα και το θέμα της ενέργειας. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται σε πολλούς κύκλους, ακαδημαϊκούς και πολιτικούς και ο πρόεδρος Μπούζεκ έχει υποστηρίξει κάποιες εργασίες, ε, σκέψεις σε αυτό το θέμα Επίσης, υπάρχουν, ε, εδώ καταλαβαίνω τις δυσκολίες διότι αν ακολουθήσουμε αυτή την κοινότητα της ενέργειας θα τίθεται το θέμα της αυτονομίας των κρατών μελών στην στρατηγική εφοδιασμού και αποθήκευσης. Είναι ένα θέμα στρατηγικής. Όλοι συμφωνούν με αυτό. Αλλά όλοι συμφωνούν επίσης ότι το επεισόδιο των συζητήσεων ανάμεσα σε ένα κράτος μέλος και την Gazprom ή τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κινητοποιήθηκε όταν υπήρχε ε, κίνδυνος μποϊκαταρίσματος από την Ουκρανία ή το θέμα ε, του τι σημαίνει ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιο, ποιος είναι ο καλύτερος αγωγός ε, αγωγός Ναμπούκο ή οποιοδήποτε άλλος αγωγός στον οποίο πρέπει να ε, δώσουμε ε, συμφωνία θα πρέπει να υπάρχει κάποια ενότητα. Γι' αυτό, σε αυτό αναφέρεται η παράγραφος 120. Θα κάνω μία πρόταση συμβιβασμού που δεν θα τηρεί απολύτως το πνεύμα της τροπολογίας που έχει υποβληθεί από το ΕΛΚ και τους φιλελεύθερους, διότι νομίζω αξίζει να το δούμε πιο προσεκτικά και ελπίζω ε, να δώσουμε μια δεύτερη σκέψη σε αυτό. Τώρα, για τα μελλοντικά διακυβεύματα της εποπτείας, πιστεύω ότι το καθήκον της Επιτροπής μας δεν είναι να ε, μπούμε στη λεπτομέρεια της νομοθεσίας, της δευτερογενούς ε, νομοθεσίας, γιατί αυτό ε, είναι σε αυτό το πνεύμα που έχω συντάξει την έκθεση και ε, που θα συντάξω και το κείμενο συμβασμού. Αλλά υπάρχει ένα σημείο όταν βλέπουμε λίγο μακροπρόθεσμα στο οποίο ε, πρέπει ανάμεσά μας εδώ να έχουμε ένα κοινό όραμα. Μια συμφωνία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Να δούμε αν θέλουμε να προχωρήσουμε προς μια αρχή, ενιαία αρχή ευρωπαϊκής εποπτείας σύμφωνα με το μοντέλο της FSA ή εάν πιστεύουμε ότι το Ολλανδικό μοντέλο Twin Peaks με μια προσέγγιση προστασίας των επενδυτών και παραγόντων της αγοράς είναι η σωστή προσέγγιση. Εγώ είμαι υπέρ της δεύτερης προσέγγισης και όχι τόσο υπέρ της πρώτης. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω δει το ισοζύγιο, την ισορροπία στην ε, ε, ε, Επιτροπή και θα πρέπει να έχουμε μια σαφέστερη άποψη. Τώρα, σχετικά με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση πρόταση 154 που είναι να αντιγραφεί ε, αυτό που έχουμε, ε, στο τομέα, έχουμε κάνει στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων υποστηρίζεται από την ομάδα των φιλελευθέρων και χαίρομαι γι' αυτό όμως είναι ένα σημείο ε, το οποίο θα πρέπει να συζητήσω με την ομάδα του ΕΛΚ διότι εκεί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία και για μένα είναι μια πολύ ισχυρή πρόταση της έκθεσης και ελπίζω να καταφέρουμε να πείσουμε τους συναδέλφους του ΕΛΚ. Την ε, παράγραφο 158 που αφορά τον πολιετή προγραμματισμό για τους εθνικούς προπολογισμούς. Αντιλαμβάνομαι ε, γιατί ενοχλεί αυτή η πρόταση γιατί μέσα στον δημοσιονομικό ε, τομέα χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις συγκυρίες. Θα πρέπει να μπορεί κανείς να διορθώνει την δημοσιονομική πολιτική ανάλογα ε, με τις συγκυρίες. Αλλά αν θέλουμε να ζητήσουμε τα κράτη-μέλη ισχυρές δεσμεύσεις και αν αυτέ οι δεσμεύσει πρέπει να είναι αξιόπιστε και το έχουμε δει στην περίπτωση τη Ελλάδα. Χρειαζόμαστε να έχουμε ε, μακροπρόθεσμα κάποιε δεσμεύσει, είτε είναι μείωση του ελλείμματο, είτε είναι χρηματοδότηση κάποιων ε, επενδύσεων που θεωρούνται στρατηγικέ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το έχουμε αυτό τον πολιτικό προγραμματισμό, διότι εμεί συζητούμε για τι δημοσιονομικέ προοπτικές αλλά μου φαίνεται ότι για μια καλή οικονομική διακυβέρνηση και μια καλή ευρωπαϊκή σύνδεση σε αυτό τον τομέα, συνάρμοση, η ιδέα του πολιετούς προγραμματισμού των προϋπολογισμών των εθνικών, χωρίς να παρεμβαίνουν ε, στο πνεύμα της επικουρικότητας, θα πρέπει να γίνει αποδεκτός. Τώρα, παράγραφος 162 είναι το θέμα των ε, δημοσίων ε, χρεών και του δημόσιου χρέους. Και είναι σημαντική αυτή η πρόταση. Ε, ίσως να πούμε να μελετήσουμε τη δυνατότητα με πιο επίο τρόπο, αλλά θέλω να αναφέρω τρία επιχειρήματα που κατά την άποψή μου είναι σημαντικά. Το πρώτο, όταν ο Επίτροπος Αλμούνια είχε κάνει τον απολογισμό των 10 ετών του ευρώ, είχε επίγνωση θέματος. Ήταν πριν από την έκρηξη της ε, κρίσης του δημόσιου χρέους, ότι ε, για ε, να προχωρήσουμε σε αυτό τον άξονα, να δώσουμε πιο πολύ δύναμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να συζητήσουμε και να δούμε τι συμβαίνει στον κάθε ευρωπαϊκό προπολογισμό. Με το Σύμφωνο Σταθερότητα έχουμε ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει ενδεχομένω ε, ε, την επιβολή κυρώσεων στο τέλο τη διαδικασία με μια, ε, ένα συνεπομισμό του χρέου σημαίνει ότι ε, ως αντάλλαγμα υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις που πρέπει να λάβουν τα κράτη-μέλη και να τηρούνται αυτές οι δεσμεύσεις. Αλλά από, άρα από πλευράς διακυβέρνησης μπορεί να είναι πολύ ισχυρό το εργαλείο αυτό. Το δεύτερο επιχείρημα και το έχουμε ακούσει όταν ε, πήγαμε στην Κίνα στην επίσκεψη. Υπάρχει μία διαθεσιμότητα κεφαλαίων σε διεθνές επίπεδο που είναι μεγάλη που ευνοεί όποια και αν είναι κατάσταση της αμερικανικής κατάστασης το, ε, την αγορά του αμερικανικού χρέους. Τώρα, αν θέλουμε ο χώρος του ευρωπαϊκού χρέους να είναι επίσης ε, ε, ελκυστικός με επιτόκια συλλογικά χαμηλά που να είναι συγκρίσιμα με τα αμερικάνικα θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό, το, αυτή την αγορά ε, στην Ευρώπη και νομίζω είναι ένα μήνυμα πολύ σαφές από το ταξίδι μας στην Κίνα. Το τρίτο επιχείρημα στο σημείο αυτό είναι η σκέψη του Προέδρου Χέρμαν Φον Ρούμπαϊ του ιδίου που σε διάφορες ανταλλαγές που είχα μαζί του λέει σε ποιο βαθμό αυτή η πρόταση του φαίνεται σημαντική και ο, ίδιος ο Πρωθυπουργός Λετέν έχει ε, ε, δώσει την άποψή του και ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ επίσης ε, και πολλοί από αυτούς που έχουν παρέμβει σε αυτό το θέμα έχουν συμφωνήσει αλλά σήμερα στην ομάδα εργασίας αυτή η πρόταση δεν έχει συζητηθεί. Νομίζω ότι η έκθεσή μας θα πρέπει να επιτρέψει το άνοιγμα αυτή τη συζήτηση σε αυτό το θέμα. Δύο σημεία, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο σχετικά με τι κυρώσει διότι υπάρχουν πολλές προτάσεις για ενίσχυση των κυρώσεων, χρήση των διαφορετικών ταμείων. Ειλικρινά πιστεύω ότι οι κυρώσεις δεν είχαν αποτέλεσμα και δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Και θέλω εδώ να αναφέρω ε, τις προτάσεις του Προεδρού Φων στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ στο οποίο συμμετείχε ένα άτυπο συμβούλιο που ε, έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα, που είπε «Ε, «Νιώθω ε, όλο και πιο άβαλα όταν βλέπω τις κυρώσεις που προτείνονται. Είναι κυρώσεις που επιδεινώνουν αυτό που θέλουμε να επιλύσουμε». Άλλες ιδέες πιο κοινωνικά ε, βάσιμες θα πρέπει να επινοηθούν. Μπορεί να θέλουμε κυρώσεις, αλλά δεν έχει νόημα να έχουμε κυρώσεις αν τι έχουμε όπως τις είχαμε στο πρώτο μέρος του Συμφώνου Σταθερότητα, γιατί δεν είχαν αποτέλεσμα. Και ε, με εκπλήττει όταν βλέπω ότι στο εσωτερικό ε, ορισμένων χωρών, μερικές φορές, η ιστορία επιτυχίας, το success story της συνοχής κάποιων χωρών είναι το πνεύμα συμμετοχής, το πνεύμα διαλόγου, η ικανότητα, δεν ξέρω στα γερμανικά υπάρχει μια μαγική λέξη, ξέρω, ε, υπάρχει μια ισχυρή συνοχή γύρω από ένα στόχο. Και αυτό ε, στηρίζεται σε ένα μηχανισμό διαλόγου πριν να υπάρχει ο μηχανισμό των κυρώσεων. Και μερικέ φορέ ε, λυπάμαι ότι σε ευρωπαϊκή επίπεδο δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτή την ικανότητα στο διάλογο, στη συνεργασία, στη συμμετοχικότητα, στη συμμετοχή πριν από την επιβολή κυρώσεων. Εάν θα υπάρχουν κυρώσει, πιστεύω ότι αυτέ οι κυρώσει θα πρέπει να είναι κυρώσει του τύπου ε, δούνου του διεθνού ε, Νομισματικού Ταμείου για να συμβάλλουν στο να γεμίσουν τα ταμεία. Είναι πιο αποτελεσματικά από το να ακυρώνονται πολιτικές που θα ήταν χρήσιμες για να συμβάλλουν στο στόχο που θέλουμε να πετύχουμε. Τελευταία λέξη για το κοινωνικό θέμα. Είναι ένα θέμα στο οποίο έχω δώσει πολύ σημασία και θα ήθελα και για κάποιες ομάδες είναι ένα θέμα δύσκολο. Εγώ θυμάμαι την ε, μετάβασή ε, μας στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας και με τους ομόλογους μας είχαμε εντοπίσει τη σημασία ακριβώς αυτού του κοινωνικού διαλόγου που αποτελεί το success story κάποιων κατών μέλων εκεί που εφαρμόζεται καλά και ε, σκέφτομαι το σκανδιναμικό μοντέλο, το γερμανικό μοντέλο για παράδειγμα. Και ε, αν κάνουμε benchmarking, γιατί να μην το μεταφέρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές τις ιστορίες επιτυχίες που παρατηρούνται σε εθνικό επίπεδο. Δεν πιστεύω ότι θα βγούμε από αυτή την κρίση χωρίς να ε, δώσουμε σημασία στην κοινωνική διάσταση που έχει προσλάβει και αυτό σε ένα συγκεκριμένο τομέα και δι τον τομέα της ενέργειας Πιστεύω δεν έχει νόημα να ε, κλείνουμε τα μάτια και να μην βλέπουμε ότι αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε συνεκτικοί στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του ε, πλανήτη, ε, είναι λογικό η ενέργεια να είναι πιο ακριβή. Αλλά αν γίνει πιο ακριβή ενέργεια, κοινωνικά είναι τρομερό αυτό το πρόβλημα, διότι όταν είστε η κυρία Μπετανκούρ, όταν είστε πάρα πολύ πλούσιος, ο λογαριασμός θέρμασης δεν είναι τίποτα. Όταν είσαι φτωχός, αυτός ο λογαριασμός είναι φρικτός, είναι αστρονομικά τα ποσά. Γι' αυτό υπάρχει ένα πρόβλημα στη μετάφραση του κειμένου, λέει η κυρία ε, Περές. Γι' αυτό μιλάω για την ασπίδα, την ενεργειακή ασπίδα που χρειαζόμαστε. Μπορεί να μην θέλουμε να προκαταλάβουμε τι θα γίνει στο κοινωνικό τομέα, αν αυξηθούν οι τιμές της ενέργειας, αλλά ε, δεν δείχνουμε ευθύνη ε, αν το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό ε, πρέπει να υπάρχει μια ασπίδα ενέργεια, μια ασπίδα στα αγγλικά η μετάφραση δεν έχει αποδοθεί σωστά. Υπάρχουν, αν το συζητήσουμε αυτό, αξίζει τον κόπο, διότι θα έχουμε μία περίπτωση όπου όλοι θα κερδίζουν. Πολύ πιο χρήσιμη. Έχω όμως ε, μιλήσει αρκετά, αλλά μερικές φορές αν έχουμε το χρόνο ε, δεν είναι κακό να αναπτύσσουμε αυτά τα επιχειρήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση. Λειτουργεί τώρα το σύστημα της ε, διερμηνίας. Ωραία, μπορώ να συνεχίσω να μιλάω γερμανικά λοιπόν. Μετά την εισαγωγή αυτή και την τοποθέτηση των βασικών ιδεών της ΠΕΒΑΣ. Θα ήθελα να καλέσω τώρα τους συναδέλφους, εάν θέλουν, να πάρουν τον λόγο. Νικόλας Χούντης, ο Λεσμίτ, Σμιτ, ποιος άλλος. Κάτσι. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε με τη σειρά των πολιτικών ομάδων και να με το ΕΛΚ, παρακαλώ. Κάτσινς. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα αγγλικά. Είχαμε πολλές, κάναμε πολλές συζητήσεις στην ομάδα μας, ε, το ΕΛΚ, για αυτή την έκθεση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πάνω από 1.600 τροπολογίες που προέρχονται από όλες τις πολιτικές ομάδες. Πράγματι, η Επιτροπή προσπάθησε να ξαναγράψει κατά κάποιο τρόπο το σχέδιο έκθεσης και συμφωνούμε με την απόφαση και τη συμφωνία της εισηγήτριας να υπάρξει μια νέα έκθεση. Να σε διακόψω. Δεν θα είναι νέα έκθεση, λέει η κυρία Μπέρες. Είναι ένα συμβιβαστικό κείμενο. Δεν πρόκειται να ξαναγράψω τα πάντα. Απλά και μόνο σας πρότεινα ένα συμβαστικό κείμενο το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τις ερωπολογίες σας. Ναι, ε, δεν θέλω ε, αυτή τη στιγμή να αρχίσουμε να διαφωνούμε ε, ε, όσον αφορά το όνομα, εντάξει. Συμβαστική έκθεση. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι μπορούμε να προσπαθούμε μπορούμε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την έκθεση αυτή, η οποία είναι ιδεολογικού περιεχομένου, ή να γράψουμε μία έκθεση, συντάξουμε μία έκθεση που να αποτελεί κοινό προβληματισμό του Κοινοβουλίου στο σύνολό του. Και εγώ σαφώς Συμφωνώ με τη στάση της εισηγήτριας που από ό,τι κατάλαβα θα καταβάλει μια προσπάθεια ε, για να συντάξει μια κοινή έκθεση με την οποία να συμφωνούμε όλοι και να μην ε, ε, εμπλακούμε σε ιδεολογικές αντιπαραθέσεις. Αυτό όσον αφορά και να σα πω τώρα και την προσωπική μου άποψη το θέμα, και εδώ είναι ιδεολογικό θέμα, δεν είναι τόσο να ρυθμίσουμε και να προστατεύσουμε, αλλά να ανοίξουμε τι αγορέ και να αγωνιστούμε για τη δημιουργία μια ε, ε, ενιαία αγορά παντού και στην ενέργεια. Με τον τρόπο αυτό θα προστατεύσουμε κυρίω του τους ε, πολίτε μα. Όχι τεχνητά δηλαδή. Να αφήσουμε τι αγορέ να ασχοληθούν με το θέμα τη προστασία των καταναλωτών. Και αυτό είναι καλύτερο για όλου. Και προτείνω σε όλου να διαβάσουν, να ξαναδιαβάσουν την έκθεση του κ. Μόντι. Και εκεί νομίζω ότι ε, υπάρχουν ιδιαίτερα ευφύεις ιδέες για το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Ε, ε, όλοι. Ευχαριστώ όλοι. Thank you very much. Well, um, Σας ευχαριστώ. Ίσως ο στόχος σας κυρία Μπέρες ήταν να μας προκαλέσετε και το καταφέρατε. Και τώρα σα ε, ξαναπετάμε το βαλάκι. Μα ακριβώ ε, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Για να συζητήσουμε όλε αυτέ τι τροπολογίε και πρέπει να σα παραδεχτώ ότι ε, εάν εδώ αρχίσαμε να κατηγορούμε ο ένα τον άλλον. Ε, πρέπει να σας πω ότι ε, εμείς ε, υποβάλαμε πολλές τροπολογίες. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο τι διαβάσατε όλες αυτέ. Ε, για να είμαστε σίγουροι ότι τι διαβάσετε, μερικέ φορέ ε, τις παραλαμβάνουμε. Ε, ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε συντονίσει καλύτερα το όλο ζήτημα. Το παραδέχομαι. Απ' την άλλη μεριά όμως και εσείς πρέπει να προσπαθήσετε ε, να ε, συντονίσετε ε, τους φιλελεύθερους και αυτό δεν είναι κάτι το εύκολο, έτσι. Τώρα, όσον αφορά το κείμενο, τη διατύπωση και ίσως αυτό ήθελε να πει και ο συνάδελφος Καρέντζη. Και πραγματικά ε, είχαμε κάποια προβλήματα. Ήταν τεράστια η δυσκολία. Αλλά καταλάβατε κι εσείς, το καταλάβατε κι εσείς ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Και προσπαθήσατε ε, ε, ε να, να καθησυχάσετε κάπως την κατάσταση. να μην εμείνουμε τώρα ιδιαίτερα στην ιστορία, παρόλο που είναι σημαντικό. Και θα έλεγα ότι ε, το να καταλαβαίνει κανεί την ιστορία είναι σημαντικό, φυσικά. Εδώ όμως ε, νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή στα σημεία στα οποία υπάρχει συμφωνία. Ανέφερα ορισμένα, αναφέραμε ορισμένα από μεριά μα ε, θέματα τα οποία πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικά. Η οικονομική διακυβέρνηση είναι ένα ε, ζωτική σημασία ζήτημα. Και θα ήθελα να σας πω ότι πριν από ένα χρόνο ορισμένοι από εμά, συμπεριλαμβάνοντα ε, και τον εαυτό μου, δεν θα παραδεχόμαστε αυτό το οποίο γίνεται σήμερα και δεν θα δεχόμαστε την πρόταση την οποία ε, κάνετε και εσείς τώρα. Παρόλο που πιστεύω ότι ε, η ομάδα του κυρίου Βαν Ρομπέη και διάβασα και τον τύπο, δεν έχει προχωρήσει όσο εμείς. Και εκείνοι λοιπόν έχουν προβλήματα. Άρα ίσως λοιπόν στο τέλος Αυγούστου θα μπορούσαμε ε, να έχουμε μια, να μας δηλαδή μια έκθεση την οποία θα μπορούσαμε και να δεχθούμε ε, σε γενικές γραμμές. Εμεί προσπαθήσαμε από μεριά φιλελευθέρων να ε, κάνουμε κάποια σχόλια. όπω ξέρετε, κατάληξαν κάποια σχόλια ε, για την έκθεση, ε, έστειλε κάποια σχόλια ε, η εισηγήτρια για την έκθεση και για τις τροπολογίες. Εμείς απαντήσαμε ε, σε 10 σελίδες, προσπαθήσαμε να τα συντονίσουμε όλα και σε επίπεδο δική μας ομάδας. Είδαμε ότι υπήρξε και κάποια διάσταση απόψεων μέσα στην δική μα την ομάδα. Μα αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Σε τελευταία ανάλυση πάντω πιστεύω ότι εμεί στην ομάδα μα θα καταλήξουμε σε μια συντονισμένη θέση και θα αντιδράσουμε ε, στις προτάσεις σας και πιστεύουμε και αυτό αν θέλετε είναι και ένα μήνυμα προς τους φίλους στην αριστερή στη δεξιά μεριά ε, ότι θα ήταν κρίμα να μην συμφωνήσουμε γενικά στο κείμενο αυτό. Δεν θέλουμε στα πλαίσια αυτά να είμαστε Ε, ε, ε, πραγματικά εμείς αυτοί που θα ψηφίσουμε σωστά. Θέλουμε όλοι να ψηφίσουμε σωστά. Είδατε τη διαδικασία ψηφοφορίας που αναλύθηκε από τον Σάιμον Τζιό από το London School of Economics που είπε ότι εμεί όσον αφορά τι ψηφοφορίε, σχεδόν στο 90% εμεί το Άλντε είμαστε στη σωστή. Ε, ε, ε από, τη, μεριά των σωστών. Εδώ δεν μα ενδιαφέρει αυτό. Γιατί αυτό που μα ενδιαφέρει και αυτό θα ήταν πραγματική προστιθέμενη αξία θα είναι ένα κοινό συμπέρασμα στο τέλο από όλου μα. Και ελπίζω όλοι να εργαστούν προ την κατεύθυνση αυτή όσον αφορά ορισμένα σημεία, σίγουρα θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά κοιτάξτε, αυτό είναι, αυτός είναι ο τρόπος εργασία μας στο Κοινοβούλιο και ελπίζω να δείξουμε αυτή την οριμότητα και στην Επιτροπή μας. Γιατί, κατά την άποψή μου, αυτό θα αποτελέσει μήνυμα για το ότι συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Αν υπάρξει ε, πολιτική κατάρρευση, ιδεολογικό πρόβλημα κτλ. τότε πραγματικά θα, υπάρξει, θα υπάρξουν δυσκολίες. Και όσον αφορά τη συνέχιση των εργασιών τη Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Μην θα σας ζητήσει τώρα το λόγο. Α, θα δώσω το λόγο πρώτα στον συνάδελφο Κάλφιν από τους σοσιαλιστές. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι εκτιμούμε την εργασία της Περβόνς. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο της. Και τώρα θα αναγκαστεί να δουλεύσει όλο το καλοκαίρι για να παρουσιάσει μια έκθεση που συνενώνει όλες τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο ανέλαβε αυτό το τόσο φιλόδοξο έργο για να έχει ένα αποτέλεσμα βέβαια και πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να είναι μια έκθεση ευρεία συνένεση στο σώμα. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα που δεν προσφέρεται για να έχουμε ιδεολογικού αγώνες, κομματικούς αγώνες. Θα πρέπει να είναι ένα σαφές κείμενο το οποίο θα πρέπει να τύχει τη υποστήριξη των μεγάλων πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω. Δεύτερον, έχοντας κατά αυτόν τον στόχο, θα πρέπει προφανώ να συμφωνήσουμε πάνω στο κείμενο. Δύο επιλογέ έχουμε. Η μία είναι να συμφωνήσουμε στο μικρότερο κοινό παρανομαστή. Σε ένα κείμενο που μπορεί εύκολα να γίνει αποδεκτό από όλους, αλλά δεν θα λέει και τίποτα. Ακολουθήσουμε αυτό που κάνει το Συμβούλιο δηλαδή και να ψηφίσουμε μια τέτοια έκθεση. Ή μπορούμε να προσπαθήσουμε το κείμενο αυτό να καλύπτει όλες τις πολιτικές ομάδες Δηλαδή όλε οι πολιτικέ ομάδε να προσπαθήσουν να κάνουν ένα βήμα προς εμπρό, έχοντα κατά νου το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πέρα τη κρίση. Και αυτό που είπε ο Σμιτ είναι ενδιαφέρον γιατί νομίζω ότι πριν από ένα-δύο χρόνια συζητάγαμε για την ε, οικονομική διακυβέρνηση κλπ. Δεν ήταν πολύ εύκολο να το συζητήσουμε. Τώρα το συζητάμε γιατί χρειάζεται και γιατί επιμένει το Συμβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε πάνω στο κείμενο αυτό και με χαρά άκουσα του συναδέλφου από τι μεγάλε πολιτικέ ομάδε ε, να παρουσιάζουν παρόμοιε απόψει. Αλλά δεν πρέπει νομίζω να χάσουμε τη φιλοδοξία να έχουμε μία έκθεση που θα παρουσιάζει μια ένα ισχυρό και ηθικό όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Έχουμε ένα εκπρόσωπο των Πρασίνων. Δεν ξέρω αν θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου. Ναι, πράγματι σε αυτή την έκθεση υπάρχουν ίσως κάποιες προκλητικές δηλώσεις, αλλά πρέπει νομίζω να είμαστε προκλητικοί, δεν μπορούμε να επανέλθουμε στα συνηθισμένα. το τελευταίο, σε εξετάζουν κάποιες αψιτροπολογίες, το θέμα του Ευρωπαίου επόπτη, πολιετή προγράμματα, Νομίζω ότι έχει δίκιο η συγγήτρια που λέει ότι αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά σημεία και δεν μπορούμε να πούμε εντάξει ας τα διαγράψουμε και ας περάσουμε στο πεπατημένο και καθημερινό γιατί ακριβώς η κρίση μας έδειξε ότι αυτό δεν είναι μια επιλογή. Χρειαζόμαστε λοιπόν προκλητική έκθεση. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Καλφέν ότι είναι σημαντικό να έχουμε συμβολή από τις πολιτικές ομάδες. Αλλά θέλουμε να έχουμε μια έκθεση ε, που θα είναι ο μικρότερο κοινό παρανομαστή, πρέπει να σταματήσουμε από τώρα. Τι να γράψουμε μια τέτοια έκθεση. Μπορεί όλοι να συμφωνήσουν, αλλά δεν θα έχει καμία, καμία επίρρεια. Γιατί όλοι ξέρουμε ποιο είναι ο μικρότερο κοινό παρανομαστή. Ε, Επίση, έχοντα κανονού το συμβασμό μετά τι θερινέ διακοπέ, θα πρέπει να ξέρουμε ότι για την οικονομική διακυβέρνηση πολλά γίνονται αυτή τη στιγμή και εξετάζουν στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Δεν χρειάζεται λοιπόν να επικαλύψουμε εμεί τι εργασίε που γίνονται εκεί. Θα πρέπει να περιοριστούμε σε εκείνα τα θέματα που μπορούν να συμβάλλουν, να προσθέσουν στοιχεία στην συζήτηση που γίνονται. Και αν ένα θέμα εξετάζεται στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, δεν χρειάζεται νομίζω να το αναπτύξουμε στη δική μα έκθεση. Επίση, η ιστορική ανάλυση είναι σημαντική, αλλά θα πρέπει να είναι πιο σύντομη γιατί θα πρέπει να ατενίσουμε το μέλλον. Και ακριβώς η μεγάλη αξία της έκθεσης είναι να εξετάσουμε πώς βλέπουμε μία ε, οικονομία εφόρο μετά την κρίση αυτή. Λοιπόν, μακροπρόθεσμα σχετικά με την πολιτική του 2020 ή τη συζήτηση για τις δημονομικές προβλέψεις ε, και προοπτικές ε, όλα το τι πρέπει να γίνει για να βγούμε από αυτή την κρίση και να έχουμε μια σταθερή και αηφόρο οικονομία. Θα πρέπει να είμαστε πιο προκλητικοί, νομίζω, γιατί βέβαια η συζήτηση γίνεται για το δημόσιο χρέος. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ιδιωτικό χρέος που εξακολουθεί να υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό. Και αυτό θα πρέπει να το αντικατοπτρίσει η συζήτησή μας. Και βέβαια αν μιλάμε για την οικονομία μακροπρόθεσμα θα πρέπει να συμφωνήσουμε και πάνω στις κοινωνικές πτυχές και συμφωνώ εδώ απόλυτα με την εισηγήτρια. Τι θα κάνουμε τελικά με την αυτή η οικονομία. Θα πρέπει να έχουμε και αποτελεσματική χρήση των πρώτων υλών. Θα πρέπει να ξέρουμε αμε, κασεκάθαρα πώς θα πρέπει να το κάνουμε αυτό γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η οικονομία θα πρέπει να είναι και ανταγωνιστική παγκόσμια και θα είναι αν κάνουμε καλή χρήση των πρώτων υλών. Ο τραπεζικό σύστημα. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς ότι χρειάζεται καλύτερο διακανονισμό, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και ποιος είναι ο τύπος του τραπεζικού συστήματος που θέλουμε Ποιε τράπεζε θέλουμε να σώσουμε και ποιε όχι, γιατί παίρνουν πολλού κινδύνου και δεν αξίζει να τι διασώσουμε με δημόσιο χρήμα. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε. Εάν δεν τα κάνουμε αυτά, θα τελειώσουμε με μια έκθεση που θα μπει κάπου σε ένα χρόνο. Έχουμε αρκετές σελίδες να εξετάσουμε, δεν χρειαζόμαστε και άλλο υλικό. Κύριε Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή. Παρόλο που είναι δύσκολη η κατάσταση, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περβόνς και εμείς ε, στην ομάδα μας θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο είναι δυνατόν. Θα θέλουμε να συνεργαστούμε. Σας αποστήλαμε τις ε, παρατηρήσεις μας και ίσως ε, τα σχόλιά μας να σας βοηθήσουμε να βρείτε συμβασμούς για την έκθεση της συμβαστική αυτή στην οποία αναφερόσαστε. Καταλήξαμε πλειοψηφικά στην άποψη που σας αποστήλαμε. Έχουμε εμπειρία από τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των πολιτικών ομάδων ε, εμπειρίες που είναι διαφορετικές και πριν και κατά διάρκεια της κρίσης. Ε, ε, βλέπουμε τώρα μια κρίση του καπιταλισμού. Ζήσαμε ήδη την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης που ήταν η κατάρρευση του σοσιαλισμού. Δεν θέλουμε να συγκρίνουμε αλλά βλέπουμε και να πούμε ότι ο καπιταλισμός έχει τα ίδια προβλήματα όπως παλιότερα η Σοβιετική Ένωση ε, ίσως δεν θα πρέπει να διατυπώσουμε τα πράγματα τόσο ομά, θα πρέπει να εξετάσουμε και τους βραχυπρόθεσμους στόχους. Δεν θα πρέπει βέβαια να προσανατολισμούμε απόλυτα στο τι κάνει το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Εμείς θα πρέπει να στοχεύουμε στους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και να αφήσουμε κατά στο το τι λέει το Συμβούλιο. Τι θα κάνουμε για την ενέργεια, πόσο λεπτομερής θα είναι η παρουσίαση στην έκθεση και θα έπρεπε η συγκήτρια να ε, πει κάτι όσον αφορά τη, την τιμή ε, της ενέργειας ή της πράσινης ενέργειας και τι γίνεται με τα μονοπόλια. Βλέπω, πούμε, τι γίνεται με την τροφοδότηση των χωρών της Βαλτικής ε, με φυσικό αέριο. Εάν δεν υπάρχει αρκετή πράσινη ενέργεια, η τιμή αυτού του τύπου ενέργειας αυξάνεται πολύ γλίγορα, έχω δει. Αλλά θα πρέπει να το εμβαθύνουμε τόσο το θέμα αυτό. Ο συνάδελφος των Πρασίρων αναφέρθηκε στο ιδιωτικό χρέος. Νομίζω ότι ο λόγος της κρίσης είναι το δημόσιο χρέος. Σε ορισμένες χώρες είναι το 100% του ΕΕΠ. Στη Λετωνία 200%, στη Μεγάλη Βρετανία 400%. Αυτά είναι τα προβλήματα. Και μέσα στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει. Άμα θέλουμε να σώσουμε την Ελλάδα ή τη Λετωνία, σώνουμε και άλλες ε, χώρες, τις τράπεζες άλλων χωρών, τα συνταξιωτικά ταμεία άλλων χωρών. Στην έκθεση δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση να αναφερθούν συγκεκριμένε προκλήσεις. Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους μετατοπίζεται στο δημόσιο χρέος και αυτό είναι κάτι που δεν αναφέρεται σωστά. Ο κ. Φαν Ρόμπε ήρθε στην ομάδα μας πριν από μερικές εβδομάδες και μας είπε ότι ο στόχος του είναι διατηρήσει τον τρόπο ζωής στην Ευρώπη. Τον ρώτησα μήπως δεν πιστεύει ότι ως πολιτικός ηγέτης θα πρέπει να δεχθεί ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, αν χρειάζονται άλλοι στόχοι για την κοινωνία. Τι σημαίνει το ε, βιωτικό επίπεδο. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε το ε, στόχο του 2020. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Άλλοι εργάζονται 35 ώρες την εβδομάδα άλλοι βγαίνουν στη σύνταξη στα 60. Ποιος θα πληρώνει όλα αυτά. Η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι στις είπα. Ε, βλέπουμε παραδείγματο χάρη είναι ε, ακίνητα που δεν μπορούν να πουληθούν παραμένουν στα, στο παθητικό τραπεζών που τα έχουν επανακτήσει. Τι σημαίνει λοιπόν ιδιωτικό επίπεδο. Εντάξει, έχουμε χρέος. Και τι, το θέμα πώς θα μπορέσουμε να εξορροπήσουμε τον προπολογισμό. Θα αυξηθεί η φορολογία. Ο Επίτροπος νομίζω δεν ασχολείται με αυτό, γιατί αυτό θα αυξήσει την ανεργία. Τι σημαίνει ευρωπαϊκό βιωτικό επίπεδο λοιπόν, τελικά. Παρόλε αυτέ τι διαφορέ, νομίζω ότι τελικά μπορούμε στην τελική έκθεση να έχουμε ένα καλό συμβασμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, η γνώμη τη ε, ομάδα μα σχετικά με το κείμενο και που έχουμε στα χέρια μα, είναι ότι είναι μια σοβαρή προσπάθεια, μια ειλικρινή προσπάθεια να ψάξει τα πράγματα και να βρει την αλήθεια και νομίζω ότι απηχεί και τον τρόπο που δούλεψε η Επιτροπή μας όλο αυτό το χρόνο, εκφράζει μια συλλογική σκέψη κτλ. Όμως η γνώμη μας είναι ότι η εισήγηση, η έκθεση, τόσο στην ανάλυση της όσο και στα συμπεράσματά της έχει ορισμένα όρια. Και πριν αναφερθώ σε αυτά κύριε Πρόεδρε και αφού μιλάμε έτσι γενικά, αν δείτε ότι ξεπερνάω το χρόνο διακόψτε με, αν είναι παραπάνω από το κανονικό της τοποθέτησή μα, επειδή θα αναφερθώ σε γενικά, διακόψτε με ε, πρόθυμο, δεν έχω κανένα πρόβλημα, επειδή θα είναι κάποιε γενικέ σκέψει. Θέλω να σα πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ε, από ό,τι αποδεικνύεται και από την προσέγγιση τη έκθεση, αλλά επειδή έχουμε το πλεονέκτημα, α το πούμε έτσι, να μιλάμε σχεδόν από του τελευταίου, ακούγοντα τι απόψει των άλλων ομάδων, κατάλαβα πάρα πολύ καλά για άλλη μια φορά ότι όταν μιλάμε για την κρίση, η οποία δεν ξέρω αν συμφωνούμε, είναι μια κρίση πολύπλευρη, όχι μόνο οικονομική, ενεργειακή, διατροφική, περιβάλλοντο ε, δεύτερο, μπορεί να είναι και πιο βαθύτερη από την κρίση του 29. Όταν μιλάμε λοιπόν για αυτό το φαινόμενο που συνέβη επί των ημερών μα, προφανώ δεν μιλάμε για ένα φυσικό φαινόμενο για την ερμηνεία του οποίου θα χρειαζόταν να επιστρατεύσουμε τις επιστημονικά, επιστημονικές, αντικειμενικές θα έλεγα, γνώσεις για να το ερμηνεύσουμε. Είναι ένα φαινόμενο που επιδέχεται ή έχει και τις αιτίες του σε πολιτικές, ιδεολογικές επιλογές και προτεραιότητε. Είναι φανερό λοιπόν ότι θα βασανιστούμε να βρεθεί συνενετικό κείμενο, καθώ όλοι μα θα επιμείνουμε ότι οι δικέ μα οι και πριν από την κρίση και στην κρίση και μετά είναι οι σωστότερε. Και αυτέ θα αποτελούσαν τη συνταγή αντιμετώπιση αυτή τη κρίση και των κρίσεων εν γέννη. Παρόλα αυτά, θα πω δύο πράγματα παρακάτω πάλι, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μία ακόμα προσπάθεια ή να συνεχίσουμε την προσπάθεια να βγει ένα κείμενο όσο γίνεται συνενετικό. Και το λέω, κύριε Πρόεδρε, από την αίσθηση ότι όσο πιο συνενετικό είναι το κείμενο που θα βγάλει η Επιτροπή τόσο θα ενισχύσει την ισχύ και την αξία του κειμένου το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι των άλλων θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέψτε μου να σας πω ότι δυστυχώς είναι υποβαθμισμένος παρά τη συνθήκη της Λισαβόνας ιδιαίτερα σε αυτά τα θέματα δεν θέλω να αφαιρθώ αναλυτικά εδώ εκπονούνται πολιτικές εδώ μιλούμε για αλλαγή συνθήκων, εδώ ε, αναφέρονται ε, στο ότι θα αυστηροποιηθεί το σύμφωνο σταθερότητα, εδώ φτιάχνονται μηχανισμοί στήριξη με τη συμμετοχή του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται κατά καιρού. Κάνουμε κάποια ερώτηση στον κύριο Μπαρόζο, παίρνουμε μια ανύπαρκτη απάντηση και συνεχίζουν τα πράγματα ω έχουν με ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρατηρητέ των εξελίξεων που είναι πάρα πολύ σοβαρέ. Επανέρχομαι όμω στην ουσία. Τα όρια που έχει το κείμενο, τα όρια που πολλέ φορέ βάζουμε στην ίδια μας τη σκέψη όσο αφορά την ερμηνεία του της δω κρίσης είναι πρώτο. κατά την άποψή μας δεν βαθύνει στις αιτίες και στις ρίζες της κρίσης που κατά τη γνώμη μας είναι αυτό που λέμε νεοφιλελεύθερο παραγωγικό καπιταλιστικό μοντέλο. Η εισηγήτρια σωστά λέει ότι αν θέλουμε να βρούμε τις απαρχές της κρίσης πρέπει να πάμε στη δεκαετία του 70 Πρέπει πράγματι να πάει στη δεκαετία του 70, τέλη της δεκαετίας του 70, μέσα της δεκαετίας του 80, όταν έχουμε επικράτηση και στο πολιτικό επίπεδο, Ηνωμένε Πολιτείε και Μεγάλη Βρετανία, ενός μοντέλου που εμπνέεται από αυτό που λέμε νεοφιλελεύθερο σύστημα. Αν δεν το δεις εκεί, η ανάλυση σου είναι επιδερμική. Διότι αυτή η συνένεση του Σουάσικτον που κυριάρχησε εν τέλει, πέρασε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συνθήκες, έχει βασικές ευθύνες για το ότι οδηγήθηκαν εδώ τα πράγματα. Και μάλιστα στηρίχτηκε με επαναπαύση ότι αυτό το μοντέλο, όπως θυμόσαστε, δεν θα ξαναφέρει ποτέ κρίση ή δεν θα ανατρέψει την ιστορία. Η ιστορία τελείωσε, τελειώσαμε. Αυτή είναι η δημοκρατία, αυτό είναι το οικονομικό μοντέλο. Όμως εδώ υπάρχουν οι διαψεύσεις των διαψεύσεων, εκτός αν κάποιος δεν θέλει να το δει. Δεύτερο, υπάρχουν προβλήματα στο ίδιο το σύστημα, αναφέρθηκε κάποιο άλλο συνάδελφο. Καπιταλιστικό σύστημα, υπάρχει πρόβλημα. Τώρα θα μου πείτε νοσταλγή σοσιαλισμού. νοσταλγώ έναν άλλον σοσιαλισμό, αλλά ε, ότι έχει πρόβλημα αυτό το σύστημα το ομολογούν και οι υπέρμαχοί του. Εδώ θέλει περισσότερο, αν θέλετε, αυτοκριτική ή κριτική διάθεση. Και τρίτο, και θα τελειώσω όσον αφορά τι γενικέ παρατηρήσει, υπάρχουν ευθύνε για την κρίση από τι πολιτικέ που ακολουθήθηκαν και σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ξαναπώ κουραστικά, κύριοι συνάδελφοι, αλλά επειδή είναι σύμφωνο σταθερότητα. Δεν έχουν γίνει τα σωστά συμπεράσματα. Η ερμηνεία που δίδεται τώρα είναι ότι χαλάρωσε, δεν το τήρησαν, δεν πειθάρχησαν ορισμένε χώρε και αυτά έφερε το αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου είναι σε λάθο κατεύθυνση. Είναι λάθο κατεύθυνση. Το ίδιο το σύμφωνο σταθερότητα είναι αντικοινωνικό, αντιαναπτυξιακό. Γιατί, α πούμε, στου όρου και στα κριτήρια που θέτει και που ετέθησαν και από τη συνθήκη του Μάστρικ, ετέθησαν μόνο το χρέο, το έλλειμμα και δεν ετέθη το ποσοστό ανεργία. Να ελέγχεται και το ποσοστό ανεργία η επιμονή στην πειθάρχηση στο σύμφωνο σταθερότητα, ενδεχομένω να διορθώσει τα δημοσιονομικά και δεν τα υποτιμώ καθόλου, αλλά θα παράξει μεγάλα κοινωνικά προβλήματα και νομίζω, χωρί να κάνω τον προφήτη, θα δημιουργήσει καινούργια κρίση. Δεν υπάρχει καμία πρόβλημα. Δεύτερη παρατήρηση είναι η ίδια η οικοδόμηση τη ΩΝΕ και του ευρώ. Κοιτάξτε τώρα τι ζούμε. Χώρε που έχουν ανάγκη να δανειστούν να μην μπορούν να δανειστούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να δανείζονται οι εμπορικέ με 1% και να βγαίνει στην ελεύθερη αγορά, να πέφτουν στα δόντια και στα νύχια των οίκων αξιολόγηση και των διάφορων κερδοσκόπων και το 1% επιτόκιο να γίνεται 5 και 6. Και δεν αναφέρουμε μόνο στην Ελλάδα, το είδατε ότι συμβαίνει και σε άλλε χώρε. Έχει δομικά λάθη. Δεύτερο, οικονομική ένωση, νομισματική ένωση, χωρί ισχυρό κοινοτικό προπολογισμό που να αναμορφώνει και να διορθώνει τι ανισοτιμίε που εξ αρχή υπάρχουν, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν είναι θα έχει προβλήματα. Και η τελευταία παρατήρηση, η λειτουργία της αγοράς. Έχουμε μια υπερδιόγκωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ακούγεται ε, ότι θα γίνει εποπτεία κτλ. Βλέπω δειλά βήματα. Εξακολουθούν να υπάρχει μεγάλη κυριαρχία. Ακόμα και τα δειλά βήματα για ε, φόρο στις ε, τράπεζες και φόρο στις τραπεζικές ε, ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές είμαστε διστακτικοί. Κατόπιν τούτου αυτή είναι η δική μα κριτική. Οι τροπολογίε μα ήταν περιορισμένε. Αν, ε, ναι, εμείς στις 1700 κάναμε 20 τροπολογίες, επιμένοντας αυτά τα σημεία προσπάθησα να σα πω. Μια τελευταία κουβέντα κύριε Πρόεδρε εδώ, μη με διακόψετε, ίσω είναι κάτι επικοδομητικό ενδεχομένως. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, ε, ρωτήσατε και σωστά τι κάνουμε τον επόμενο χρόνο. Τι κάνουμε τον επόμενο χρόνο. Ε, θα έλεγα να συνεχίσουμε την προσπάθεια να, να τελειώσουμε τη δουλειά μα αν είναι δυνατόν να υποθεί αυτή η λέξη και ας απασχοληθούμε τον επόμενο χρόνο, εμένα θα μου άρεσε προσωπικά, πώς αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις εν γέννη, δηλαδή να μην μας ξανασυμβεί, αν μπορούσαμε να πούμε κάτι. Και εκεί βέβαια θα έχουμε τις διαφορές μας, αλλά ας γράψουμε, εγγράψουμε ο καθένας για την ιστορία τι προέβλεψε και τι δεν προέβλεψε. Θα έχει, μια, θα ένα δημιουργικό χαρακτήρα μια τέτοια προσπάθεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τρεις ε, συνάδελφοι έχω ακόμα Μπότας, η αντιπρόεδρά μας και με ο απευθυνόμενος μετά. Καταρχήν χαίρομαι που επανήλθε ο Μικέλ, ήταν άρρωστος αρκετές εβδομάδες και γι' αυτό απουσίαζε. Καλώς ορίσατε λοιπόν πάλι, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω μία ε, ε, ε παρέμβαση, η οποία βέβαια δεν θα είναι τόσο λεπτομερή όσο ο προηγούμενο συνάδελφο, αλλά έχει να κάνει με ένα σχόλιο του συναδέλφου από το ΕΛΚ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει ε, ναι, ε, αναφέρθηκε στο ιδεολογικό ζήτημα ε, και στο γεγονό ότι πρέπει να αφήσουμε τι ιδεολογικέ ε, ε αντιπαραθέσει. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμένα ε, μου φέρνει στο μυαλό αυτό το πίνακο του Μαγκρίτ με τίτλο «Σε είναι Πάζιν πίπ, ότι αυτό δεν είναι μία πίπα. Μα κοιτάξτε, ήταν δηλαδή αυτό δείχνει, αλλά δεν θέλει να αναφερθεί σε αυτό. Ε, μα κοιτάξτε, τελικά η ιδεολογία μένει πίσω από τον πίνακα. Και όχι εδώ ε, το θέμα δεν είναι να μιλάμε για την πραγματικότητα, να τη βλέπουμε όμω ταυτόχρονα την πραγματικότητα. Αυτό ο πίνακα λοιπόν, του Μαγκρίτη είναι καθαρά ιδεολογικό. Και νομίζω ότι θα πρέπει να εργαστούμε ιδιαίτερα, να εργαστούμε πάρα πολύ. Και κυρίω, ε, ε, ε, η κυρία Μπερέ, ε, όσον αφορά τις τροπολογίες αυτές των 1600 και, και βάλε, εμείς ε, ε, παρουσιάσαμε 20 τροπολογίες. Ε, αλλά όλοι μας θα πρέπει να δούμε τα επιχειρήματα, τι επιχειρήματα θα χρησιμοποιήσουμε και τι επιχειρήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Όταν κάποιο λέει, α αφήσουμε τη βιολογία εκτός της έκθεσης, Λοιπόν, τι μου έρχεται στο μυαλό. Μα τι μου έρχεται. Αυτή η πρόταση τελικά είναι ιδεολογική πρόταση, δεν είναι. Και μάλιστα να σα πω ότι πριν από ένα χρόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε 440 εκατομμύρια ευρώ στην τραπεζική τράπεζα και τώρα ε, στην αγορά ε, και το, με 1%. Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται, πρέπει να πληρωθεί αυτό το ποστό. Ε, τι έγινε στο μεταξύ. Στο μεταξύ, με αυτά τα χρήματα, ορισμένε από αυτέ τις τράπεζε αυτό που έκαναν ε, είναι να αγοράσουν κρατικά ομόλογα. Ε, τότε μιλάγαμε για 3%. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προτείνει ε, να, να, δούμε την, να, να οργανώσει την αγορά αυτή των ομολόγων. Ναι, ενδιαφέρουσα ε, είναι αυτή η πρόταση, αλλά πώς αγοράζονται από τι τράπεζε με 4 και 5%. Ε, μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ μπορούμε να δούμε το θέμα κάτω από δύο σκοπιέ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, διασώζει το τραπεζικό σύστημα, σωστό, αλλά και κάτι άλλο που με ενδιαφέρει περισσότερο εμένα. Ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ε, χαζή ή τελικά τι κάνει. Ε, σώζει ε, ε τα δημόσια οικονομικά. Γιατί τι κάνει στην ουσία. Χρηματοδοτεί με τον τρόπο αυτό. Γιατί ε, ε, προτείνει χαμηλά και τελικά αγοράζει ακριβά. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, ανάλογα με την ανάλυση χρησιμοποιούμε και τα ανάλογα επιχειρήματα. Αλλά να σας πω ότι ε, πρέπει να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε επιχειρήματα ε, που, και να λέμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε επιχειρήματα που τελικά έχουν να κάνουν με την ουσία του ζητήματος. Αυτό ήθελα να πω, Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Kiitos on helppo jatkaa Karl Marxia, koska hän sanoi, että... ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο Καρμάξ είπε ότι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση είναι πιο σημαντικό από μια ντουζίνα σωστά προγράμματα. Υπάρχουν πολλές προτάσεις στο πώς θα ξεπεράσουμε την κρίση. Η έλλειψη εμπιστοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντική εδώ στην Ευρώπη. Ακούσαμε διάφορους εμπειρογνώμονες ε, όταν τους είχαμε καλέσει εδώ. <clears throat> Πολλοί εμπειρογνώμονε είπαν ε, ότι θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε την κρίση παραδείγματο χάρη με το ε, βόρειο πρότυπο, σκανδιναβικό πρότυπο. Αυτό τι σημαίνει πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Θα πρέπει να δούμε προς ποια κατεύθυνση κινούμεθα. Εμείς στην Ευρώπη δεν έχουμε την εμπιστοσύνη που χρειαζόμαστε. Εμπιστοσύνη χρειάζονται όλοι. Θα πρέπει να μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις κατά πόσο θέλουμε να δημιουργήσουμε πραγματικά εμπιστοσύνη με τη δική μας εργασία. Ή όχι, νομίζω ότι όλοι θέλουμε να επανέλθουμε σε μια κατάσταση εμπιστοσύνης. Και αυτό είναι σημαντικό η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Και θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στις προτεραιότητες, στα σημαντικά θέματα. Χρειαζόμαστε συνένεση, χρειαζόμαστε να κινηθούμε προς την ίδια κατεύθυνση. Και νομίζω ότι αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Όπω είπε εισαγωγικά και η Περβόνς το το πυρήνα του προβλήματο είναι ότι παραδείγματο χάρη στο ΕΛΚ όταν εξετάζει κανένα τις τροπολογίε, βλέπει ότι υπάρχουν περισσότερες διαφορέ στο εσωτερικό του ΕΛΚ από ότι μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Και απόρρισα που είπε ο εκπρόσωπος του ΕΛΚ ότι ε, στην ενεργειακή πολιτική δεν είναι σημαντικό ο καταναλωτής και ο φιλοδός μου συνάδελφος εδώ βλέπω ότι έγνεψε καταφατικά. Μα δεν πρέπει να ξεχνάμε ποια είναι η κεντρική ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε αξίες, ε, χρειαζόμαστε κοινά προγράμματα, χρειαζόμαστε και τους καταναλωτές όμως. Αυτή είναι η ιδέα. Λοιπόν, Καλή είναι η ιδεολογία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, έχουμε μία κομματική ιδεολογία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για την αντιμετώπιση της κρίσης πρέπει να έχουμε κατά νου την ίδια την ιδέα, την ίδια την ύπαρξη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν αξιολογηθεί αργότερα η απόδοσή μας θα δοθεί σημαντική, σημαντικό βάρος στον τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο αντιμετώπισε την κρίση αυτή. Ε, το θέμα της εποπτείας δεν είναι πολύ καλό παράδειγμα μου φαίνεται. Ούτε θα ήταν καλό βέβαια να ψηφίσουμε πάνω στις 1600 ε, τόσες τροπολογίες χωριστά. Θα πρέπει να αντιστοιχθούμε τολμηροί. Πρόεδρο, που του δώσα το λόγο στην Περβόνς για να ολοκληρώσει, θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω όλα αυτά που ελέγχθησαν, αλλά θα ήθελα πώς να παρατηρήσω ότι εμείς ως Επιτροπή έχουμε την ευκαιρία το Σεπτέμβριο να πετύχουμε μεγάλη ε, ομοφωνία πάνω στην έκθεση και έτσι να μπορούμε να έχουμε σημαντικό λέγειν πάνω στη συζήτηση που έχει ξεκινήσει η ομάδα Φανερών Πόη είναι ένας παράγοντος η Κομισιόν έτσι και αλλιώς καλείται να τοποθετηθεί και εκείνη και το Κοινοβούλιο με μια τολμηρή έκθεση η οποία θα τύχει τη συνένεση της πλειοψηφίας μπορεί πραγματικά να εισακουστεί. Και γι' αυτό είναι σημαντική και χρονική στιγμή κατά την οποία θα ολοκληρώσουμε. Θα πρέπει το Σεπτέμβριο να είμαστε έτοιμοι. Θα πρέπει μέχρι αρχές ή μέσα Σεπτεμβρίου να καταλήξουμε να έχουμε συνένεση. Ακόμα και αν δεν έχουμε ψηφίσει, θα μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο να παρουσιαστούμε στην κοινή γνώμη με τις απόψεις μας. Ένα αυτό. Δεύτερον, στην τελευταία ανάλυση νομίζω ότι είδαμε ότι έχουμε μια ηθική και μια πολιτική κρίση. Η πολιτική κρίση αναφέρθηκε πριστάκι όσον αφορά την Ευρώπη. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως κάναμε μέχρι στιγμής. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ τολμηρές απαιτήσει. Ακόμα και αν ξέρουμε ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν σήμερα ή αύριο. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη Ευρώπη σε πολλού τομεί από εκείνη που έχουμε σήμερα. Αυτό δεν αρέσει τα κράτη-μέλη γιατί ε, στην κυριαρχία του, στην ανεξαρτησία του κλπ. Αλλά αυτό είναι όμω γεγονό. Το είδαμε από τι εξελίσσει ότι σε πολλού τομεί ενέργεια ένα από αυτού αλλά και άλλου, σε πολλού τομεί λέω χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και θα πρέπει να το πούμε Ξεκάθαρα. Κατόπιν έχουμε μια ηθική κρίση που δεν θα μπορέσουμε και τόσο πολλά να κάνουμε βράχη πρόθεσμα γιατί πολλές από τις αξίες οι οποίες ίσιαν μέχρι στιγμής χάθηκαν τα τελευταία χρόνια τις τελευταίες δεκαετίες και δεν νομίζω ότι υπάρχει τόση πολύ βούληση για αλλαγές αλλά και κοιτάξω όλο τον χρηματοπιστωτικό τομέα Βλέπω ότι πολλοί πέρασαν στο business as usual, στα πεπατημένα. Και βλέπουμε ότι η μεταρρύθμιση της ΕΠΑ δεν έχει υπογραφεί, δεν έχει περάσει στην νομοθεσία και ήδη, ήδη οι ενδιαφερόμενοι βρίσκουν τα παραθυράκια που θα τους βοηθήσουν να ε, υποσκάψουν αυτά που έχουν αποφασιστεί. Λοιπόν, έτσι δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Αλλά όσον αφορά την πολιτική κρίση, ιδίω την πολιτική κρίση στην Ευρώπη, μπορούμε νομίζω να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και εκεί θα πρέπει νομίζω να βρούμε μια λύση που θα ξεπερνάει τα όρια των κομμάτων και των πολιτικών ομάδων. Μετά κάποιο αναφέρθηκε στο θέμα ότι δεν πρέπει να επικαλύψουμε τι εργασίε μα με τι εργασίε άλλων επιτροπών, παραδείγματο χάρη τη Επιτροπή ΕΚΟΝ. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δεν θα πρέπει να αναφερθούμε στο θέμα τη εποπτεία. Δεν χρειάζεται να μπούμε στι λεπτομέρειε. Αλλά θα πρέπει παρόλα αυτά να πούμε ξεκάθαρα ποιε είναι οι απόψει που προσπίζουμε εδώ, για να είναι σαφέ ότι εδώ το Κοινοβούλιο είναι ενωμένο στην άποψη αυτή πέρα από τα, τις μεμονωμένες επιτροπές να πούμε ότι προτιθέμεθα να δεχτούμε περισσότερη Ευρώπη και λιγότερη κρατική παρέμβαση. Αυτά είχα να πω, τον τελευταίο λόγο έχει υπερβόνς και μετά μπορούμε να κλείσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την ε, συνάντηση διότι αυτό με ενθαρρύνει. Με ενθαρρύνει πολύ στο, σε αυτή την πρόκληση που ε, έχω προτείνει να ε, υποβάλουμε ένα συμβαστικό κείμενο επιτάπητος. Ο συνάδελφος Κάριντς έχει φύγει, αλλά ε, δεν είμαι εχθρική προς τις αγορές, αλλά σας λέω, ως εισηγήτρια ε, εγώ, πιστεύω ότι οι καλύτεροι υπερασπιστές των αγορών είναι οι σοσιαλιστές, διότι γνωρίζουν ότι μια αγορά χρειάζεται ρύθμιση και όταν οι σοσιαλιστές ε, αποδεχτούν τη λειτουργία μιας αγοράς είναι οι καλύτεροι υπερασπιστές. Δεν θέλω αυτό να βάλω όμως στο συμβιβαστικό μας κείμενο. Ε, αυτό που θέλω να πω στους έναν είναι ας πάρουμε τον τομέα της ενέργειας για παράδειγμα γνωρίζουμε ότι είναι ένας πολύ καπιταλιστικός τομέας όπου οι στατικικές επενδύσεων, μακροπρόθεσμων επενδύσεων είναι απαραίτητες και βλέπουμε πολύ καλά ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί απλά να είναι ένας ρόλος ε, όπου ε, θεσπίζονται κανόνες της αγοράς. Εμένα πάντα με εκπλήττει, γιατί ε, θαυμάζω μάλλον αυτό που έγινε υπό την Γερμανική ε, Προεδρία το Μάρτιο του 2007, διότι είχαμε θέσει του κανονισμού σε ό,τι αφορά την ενέργεια και τι κλιματικέ αλλαγέ. Αλλά με απογοητεύει αυτό που κάναμε, διότι τελικά κάναμε ένα πρόβλημα εσωτερική αγορά. Ναι, υπάρχει πρόβλημα εσωτερική αγορά, αλλά δεν υπάρχει απλά πρόβλημα εσωτερική αγορά. Υπάρχει και πρόβλημα έρευνα, ανάπτυξης, οράματος, ε, μακροπρόθεσμων επενδύσεων πολύ ωραία για τον τομέα της ε, αγοράς της ενέργειας, αλλά δεν αρκεί αυτό. Σε ό,τι αφορά την έκθεση Μόντι, συμφωνώ. στι τροπολογίε που έχω συνθέσει, έχω προσθέσει από την έκθεση Μόντι, όμως η έκθεση Μόντι είναι ε, σε, μια, σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν πρέπει να ε, ξεχάσουμε στα θέματα οι εκπρόσωποι έχουν αποχωρήσει όμως από την ε, αίθουσα σχετικά με το δημοσιονομικό θέμα. Ευχαριστώ τον Όλε Σμιτ. Αν τον έχω προκαλέσει, πρέπει να σας πω Συνάδελφε, με γνωρίζετε εδώ και αρκετό καιρό για να ξέρετε ότι αν μου έχετε εμπιστευτεί αυτή την έκθεση δεν είναι για να σας κάνω κάτι ε, το μη... Ε, σας έχω κάνει κάτι πολύ σοβαρό. Χαίρομαι που σας έχω επιτρέψει, που σας έχω υποχρεώσει να δουλέψετε για να επανισορροπήσουμε τα πράγματα. Αλλά έχω βάλει αυτά που στεύω εγώ ως εισηγήτρια και έχω πείγνωση του θέματος ότι ε, μπορεί να μην ε, είναι η κοινή άποψη όλων. Γι' αυτό ε, προτείνω να υποβάλουμε τώρα ένα συμβαστικό κείμενο. Αν με επιτρέψετε, δεν θα ακολουθήσω το να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε τους φιλελεύθερες, διότι εγώ θα προσπαθήσω να συντονίσω όλους. Είναι ακόμη πιο φιλόδοξο έργο αυτό, αλλά εμπίπτει περισσότερο στην εντολή μου. Και σας αφήνω εσάς ε, να συντονίσετε τους φιλελεύθερους. Και συμμερίζομαι την άποψή σας ότι θα κερδίσουμε εάν συγκεντρωθούμε στο μήνυμα ακριβώς ε, ε, και ξέρετε υπάρχει πολύ καλή ο συντονισμός με τον Πρόεδρο που ανήκει και στην ομάδα σας αν συγκεντρωθούμε στο ισχυρό μήνυμα το οποίο θέλουμε να μεταδώσουμε προς τα έξω. Και απαντώ και στον Πρόεδρο λέγοντας ότι ε, στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων υπήρχε, υπήρχαν κάποια ερωτηματικά. Αλλά υπάρχει κρίση, δεν πρέπει να δώσουμε άμεσες απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών. Και ε, είπαμε δεν θα ικανοποιήσουμε τίποτα με αυτές τις άμεσες απαντήσεις. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρίξουμε φως, να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα για το μακροπρόθεσμο όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα βρούμε κάποια συνένεση και θα δούμε ποιο είναι ο ρόλος αυτής της έκθεσης τελικά. Είπατε ότι πρέπει να εστιαστούμε πολύ στην ιστορία, υπερβολικά στην ιστορία. Με πλήττει αυτό, διότι όταν είχαμε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είδαμε ότι εκεί ε, κινούνται προ ένα νομοθετικό πακέτο, αλλά δεν είχαν συμφωνήσει για τα αίτια της κρίση. Και εδώ τα πράγματα είναι λίγο πολύ τα ίδια. Δεν το λέμε ανοιχτά, αλλά κάποια σημεία της ανάλυση των αιτίων της κρίση εκεί υπάρχουν διαφωνίε. Και θα παραμείνουν και πέραν από αυτή την έκθεση που ε, θα υιοθετήσουμε, θα εγκρίνουμε τον Οκτώβριο αυτό που μπορούμε να δούμε στην κοινή ανάλυση των αιτίων θα πρέπει να το εντάξουμε στο κείμενο, αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν θα είναι εξαντλητική ανάλυση αυτή. Συμφωνώ απόλυτα με τον ε, συνάδελφο Ιμποκελφάν και θα ακολουθήσω τις ε, ε, συμβουλές του και θα πάω θα ακολουθήσω τις συμβουλές του, αλλά μου φαίνεται ότι ε, αυτό είναι και βούληση ε, άλλων ε, συναδέλφων. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα του, της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Η δευτερογενής ζητομοθεσία δεν είναι δικό μας θέμα και δεν είναι δική μας δουλειά. Υπάρχουν δύο θέματα στα οποία δεν μπορούμε να παραμείνουμε αμήλυτοι και το πρώτο είναι η οικονομική διακυβέρνηση όπου στην ε, ΕΚΟΝ ε, υπάρχει μια έκθεση που θα κάνει ο κύριος Φέγιο και εγώ θέλω και ελπίζω να, ε, ελπίζω να συμφωνούν οι συνάδελφοι να συντονιστώ μαζί μου διότι δεν μπορούμε σε αυτή την έκθεση να μην αναφέρουμε τίποτα για την οικονομική διακυβέρνηση. Είναι αδύνατο να μην αναφερθεί τίποτα και είναι δίκαιο και η Επιτροπή ΕΚΟΝ να αντιδράσει σε αυτό το θέμα. Αλλά εκεί χρειάζεται πραγματικά να υπάρχει μία παράλληλη προσέγγιση. Και ίσως στην Ολομέλεια, όταν θα συζητήσουμε την έκθεσή μας, η έκθεση του κύριου Φεγιό μπορεί να ε, συνδυαστεί στη συζήτηση. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό, αλλά θα πρέπει να έχουμε αυτή την προσέγγιση. Τώρα, στο θέμα της εποπτείας, τα πράγματα είναι λιγότερο περίπλοκα, διότι και στην Επιτροπή ΕΚΟΝ ε, βλέπουμε κείμενο προς κείμενο και ε, δεν είναι μια σφαιρική άποψη και τα σημεία τα οποία βλέπουμε εμείς στην έκθεσή μας είναι θέματα που δεν ε, είναι ε, θέματα συζήτηση, είναι μακροπρόθεσμα. Ο κύριος Τσίλε έχει αποχωρήσει. Όχι, είναι εδώ, είναι εδώ ακόμη μαζί μας. Το απαντάω λοιπόν αμέσως. Αυτό που είπατε για το σοβιετικό σύστημα και το κεφάλαιο κίνησης είναι συγκινητικό, διότι αυτό που μαθαίνουμε στο Κοινοβούλιο είναι ότι ο καθένας έχει διαφορετική, μια διαφορετική ιστορία πίσω του. Και εμείς θα πρέπει να συνδυάσουμε αυτές όλες τις ιστορίες. Και σας διαβεβαιώ ότι αυτό, αυτή τη στιγμή δεν έχω εναλλακτικό σύστημα. Αλλά θέλω να λειτουργεί σωστά ο καπιταλισμός και θα πρέπει να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία και όχι τους θεροσκόπους. Ε, δεν πρέπει να ε, δανειζόμαστε λεφτά για να βγάζουμε λεφτά, αλλά για να χρηματοδοτήσουμε την πραγματική οικονομία. Και είναι αυτό ίσως που ε, ξεχάστηκε από τους ε, ε, κακούς δημιουργούς του καπιταλισμού. Ευχαριστώ που συμφωνείτε ότι δεν πρέπει να εστιαστούμε στην καθημερινή εργασία του Συμβουλίου. Τώρα στο θέμα του δημόσιου χρέους. Παράγραφος 17 λέει ρητός ότι αυτή η κρίση έχει οδηγήσει σε μια μεταφορά της του ιδιωτικού χρέους σε ένα δημόσιο χρέος. Λέτε ότι δεν είναι σωστά ανεπτυγμένο, αρκετά ανεπτυγμένο και βλέπω την ε, τροπολογία 218 που έχετε υποβάλει, αλλά δεν την έχω ε, ακολουθήσει στην ακαιρεότητα διότι υπάρχει μόνο μία ε, πτυχή ε, του θέματος. Το θέμα της μεταφοράς του χρέους σε δημόσιο χρέο δεν είναι μόνο πρόβλημα των νέων κρατών μελών, είναι και πρόβλημα των οικοκυριών ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι ένα πιο παγκόσμιο πρόβλημα. Φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο το προσεγγίζεται. Ίσως να πρέπει να βρούμε μια φόρμουλα έτσι ώστε να ε, γίνει πιο ε, ρητός εκπεφρασμένο αυτό το ε, σημείο. Και να συνοψίσεις καλά την κατάσταση. Ο κύριος Σκουντής, όταν λέτε ότι στο σύμφωνο σταθερότητα δεν τη χειρισμού το θέμα της απασχόλησης και ότι είναι ένα από τα λάθη αυτού του συμφώνου. Συμφωνώ 100% με αυτήν την άποψη. Το είπα και στον πρόεδρο Χέρμαν Φαν και είναι ένας από τους φόβους που έχω για τη λειτουργία αυτής της ομάδας εργασίας. Όταν νομίζουμε ότι η διακυβέρνηση οικονομική θα λυθεί μόνο από τις υπουργού ε, οικονομικών, δεν είναι η σωστή ισορροπία αλλά ε, υπάρχει ε, το, επίγον της, ε, της υπόθεσης εδώ. Κύριε Πόρτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμβουλές σας. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο. Κύριε Γιακοντσαρή, σας ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις γιατί αγγίζουν πραγματικά την ουσία του έργου μας. Και παραπέμπουν σε αυτό που είπα για το σκανδιναβικό ή το γερμανικό μοντέλο προηγουμένως. και επίσης την ε, κατάσταση στην Ελλάδα. Ένας Αμερικανικός συνάδελφος ε, μου το ανέφερε αυτό το Σαββατοκύριακο. Μία από τις δυσκολίες της ε, ελληνικής κοινωνίας είναι μια κοινωνία όπου υπάρχουν πολλές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Ε, δεν θέλω βέβαια να αγκαλιαζόμαστε όλοι και να αγαπιόμαστε, αλλά σε αυτόν τον περίπλοκο κόσμο που ζούμε, οι κοινωνίε όπου υπάρχει ένα βαθμό εμπιστοσύνη και μια ικανότητα εμπιστοσύνη ε, ε, και συνεργασία, στο σύγχρονο κόσμο και στην κατάσταση όπου βρισκόμαστε σήμερα στην Ευρώπη ε, απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, αυτές οι, οι κοινωνίες θα βγάζουν πέρα καλύτερα και ε, θα πρέπει να δώσουμε στην Ευρώπη αυτή τη δυνατότητα και είναι οι προτάσεις που κάνουμε στην έκθεση αυτή που θα συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Πρόεδρε, τις επιθυμίες σας όταν λέτε ότι ως Επιτροπή Κρίσης έχουμε μεγάλη ευκαιρία να ε, υποβάλουμε αυτή την έκθεση, αλλά λυπάμαι ότι ε, οι περισσότεροι οι συνάδελφοι δεν συμμερίζονται το θέμα ότι αυτή η κρίση είναι η κρίση ηθική και πολιτική, όπως ξέρετε στην παράγραφο 22, το έχω πει ρητός όταν πήγαμε στη Νέα Υόρκη, ε, μας ε, μας φιλοξένησε το, η Οξφόρδη των αναλυτών που χαιρέτησαν αυτή την πρόταση ως μια πολύ ισχυρή πρόταση αυτής της έκθεσης αλλά βλέπω ότι δεν ε, συμμερίζονται ε, μια, πολιτική, μια πολιτική ομάδα δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη και δύο μέλη έχουν προτείνει την διαγραφή αυτής της αναφοράς αλλά στο συμβαστικό κείμενο σας διαβεβαιώ ότι θα λάβουμε υπόψη κάποιες προτάσεις και, και θα μείνει στην έκθεση. Ωραία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν. Και ραντεβού όταν επιστρέψουμε από τις θερινές διακοπές για να βάλουμε τις τελευταίες πινελιές. Σας ευχαριστώ όλους για τις συμβουλές. Σας ευχαριστώ την Περβόνς. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση και ελπίζω να σας δω όλους αρχές Αυγούστου, ε, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου.